Der Präsident! Die Sitzung ist wieder auf. Ε, άρχεται η συνεδρίαση. Η κυρία Φιγκερέντο ε, έχει ένα, ένα διαδικαστικό επί της ημερησίας διατάξεως. Κύριε Πρόεδρε, είναι ένα διαδικαστικό λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα το πρωί είχαμε εδώ ψήφο